Habt ihr mich alle verstanden? Gut. Ich bin noch im Amt, bis die neue Vorsitzende... Με ακούτε όλοι? Λοιπόν. Κυρίσω την έναρξη της συνεδρίασης. Το επόμενο βήμα είναι η εκλογή του Πρόεδρου της Επιτροπής μας. Πρέπει να εκλεγεί πρόεδρος, τέσσερις αναπληρωτές, ε, δηλαδή τέσσερις αντιπρόεδροι. Καταρχήν να δούμε αν έχουμε απαρτία. Χρειάζονται 8 τουλάχιστον μέλη και είναι φανερό ότι έχουμε την απαρτία. Για την Προεδρία. Από το ΕΛΚ υποψήφια η Doris Πακ. Εγώ ίδια δηλαδή. Ξέρω ότι η ομάδα μου με πρότεινε. Ελπίζω ότι το κάνανε με πεποίθηση κιόλας. και επομένως συμφωνώ να είμαι υποψήφια. Η δήλωση οικονομικών συμφερόντων δεν έχουν αλλάξει, είναι αυτά τα οποία θα βρείτε και στο διαδίκτυο. Μπορεί να γίνει λοιπόν η ψηφοφορία διαβοής ή με μυστική ψηφοφορία, εάν κάποιος το επιθυμεί. Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε. Α, σας ευχαριστώ. Στον πρώτο γύρο η Ντόρις Πάκα έχει εκλεγεί πλημμυρίζω από συγκίνηση. Θα ήθελα λοιπόν δι, να, ή σηκώνει ανατάσεως χειρών να εκλέξετε την Doris Πακ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε ξεπεράσει λοιπόν τον Ποτοσκόπελο. Έχω επανεκλεγεί, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ελπίζω ότι θα είμαι στο ύψος των προσδοκιών σας και ότι θα είμαι λιγότερο πιεστική και λιγότερο κουραστική σε αυτό το δεύτερο γύρο. Θα κάνω προσπάθεια να είμαι λίγο πιο αγαπητή σε εσά και λίγο πιο αυρόφρονα. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και θα το συνεχίσω αυτό. Αντιπρόεδρε. Τέσσερι προτάσει για αντιπροέδρου. Η πρώτη πρόταση, η κυρία Χέλγα Τρίπελ από του πράσινου Εάν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, όλα αυτά τα οποία ρωτήσατε για μένα ισχύουν και για μένα. Έχει συμφωνήσει η κυρία Τρίμπελ, έχει κάνει όπως έπρεπε τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων, την έχει προτείνει η ομάδα της, δέχεται την ε, πρόταση αυτή. Όποιος είναι υπέρ της κυρίας Τρίμπελ μπορεί να την εκλέξει δια voice ή δια χειροκροτημάτων. Πολύ ωραία. Μπορείς να έρθεις και στα θεωρία του Προεδρείου, στις θέσεις του Πρόεδρου. Η δεύτερη θέση Πρόεδρου. Πρόκειται από την ομάδα για την ελευθερία και την δημοκρατία που έχει μια νέα πρόταση έναν Ιταλό συνάδελφο, τον κύριο Φοντάνα. Κύριε Φοντάνα, θέλετε να πείτε κάτι για τον εαυτό σας, για το άτομό σας, για να γίνετε πιο γνωστό στην Επιτροπή μας. Κύριε Φοντάνα, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να πω ότι έως σήμερα εργαζόμουν στην Επιτροπή Αλίας, όπως και επιφαλής της ομάδας μου. Κάναμε εξαιρετική δουλειά με τον πρόεδρο Τεκάστρο. Ακριβώς επειδή εργαστήκα πάνω στο θέμα της κοινή αλληλευτικής πολιτικής από τα πλέον σημαντικά ζητήματα, τώρα έχω τη δυνατότητα να συμμετάσχω σε εργασίες Επιτροπής Πολιτισμού. Ήταν η, Επιτροπή προτιμούσε αυτής εξ αρχής, οπότε χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι μαζί σας. Ελπίζω να με καλοδεχτείτε στην Επιτροπή σας εξίσου καλά όπως οι συνάδελφοι στην Επιτροπή Αλίας και ελπίζω να έχω μια επικοδομητική σχέση με όλους. Σας ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο η πρόεδρος. Ευχαριστώ λέει κύριε Φοντάνα και συνεχίζει πάλι χωρίς μικρόφωνο. Η ψυχή της Ευρώπης δεν βρίσκεται στην Επιτροπή Γεωργίας αλλά στην Επιτροπή Κουλτούρας, Πολιτισμού. Χαιρόμαστε που είσαστε μαζί Όποιο είναι υπέρ του κύριου Φολτάνα, παρακαλώ να δείξει τη θέση του με χειροκροτήματα. Ευχαριστώ. Μπορείτε να έρθετε κι εσείς, αγαπητέ συνάδελφε. Τρίτη πρόταση. Θέση τρίτου αντιπρόεδρου από την ομάδα της αριστεράς. Ο κύριος Μπίσκι, δυστυχώς είναι άρρωστος ο κύριος Λόταρ Μπίσκι, αλλά έχει αποδεχθεί την υποψηφιότητα αυτή. Έχει κάνει όλα τα άλλα απαραίτητα διαβήματα και σας προτείνω εφόσον τον υποστηρίζει και η ομάδα των αριστερών, να τον δεχτείτε και αυτόν με χειροκροτήματα. Ευχαριστώ. Δώστε τα χαιρετίσματά μα στον κύριο Μπίσχη και ευχέ για ταχεία ανάρρωση. Τελευταίος αντιπρόεδρος από τους φιλελεύθερου, ο Μάρτιν Κλόπεγκάτ, ο οποίος και αυτό έχει κάνει τι απαραίτητε ενέργειε εφόσον η υπομοιδιά είναι σίγουρο ότι τα έχει πράξει. Θα ήθελα λοιπόν να επιβεβαιώσετε και τη δική του εκλογή. Σας ευχαριστώ. Ελάτε κι εσείς και έχουμε εκλέξει το, το νέο Προεδρείο της Επιτροπής μας. Εύχομαι σε όλους καλή συνεργασία στα δυόμιση χρόνια που μας περιμένουν. γιατί θα έχουμε πολύ σημαντικά θέματα να αντιμετωπίσουμε, τα πιο σημαντικά ίσω θέματα που έχει ποτέ χρειαστεί να αντιμετωπίσει η Επιτροπή Πολιτισμού. Μπαίνω τώρα στα κύρια θέματα της ημερησίας διάταξης. Έχουμε καταρχήν την έγκριση της ημερησίας διάταξης, αν δεν υπάρξει καμία αντίρρηση. <clears throat> Μπορούμε να συνεχίσουμε με την προτινόμενη ημερησία διάταξη. Ανακοινώσει τη Προέδρου. Δεν έχουμε τσεχικά, εστονικά, λιθουανικά, λετονικά, λετονικά, εστονικά, σλοβενικά, ούτε και σουηδικά. Αυτές οι γλώσσες μας λείπουν. Όλες οι άλλες είναι παρούσες. 4. Σημείο 4. Επιγραμμική διανομή διανομή όπτικο-ακουστικών έργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η συγγυσία του κυρίου Καβαντά. Κύριε Καβαντά, έχουμε κάνει μια πρώτη συζήτηση για αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να παρουσιάσετε και πάλι μαζί με τα σχόλιά σας την ε, έκθεση αυτή πρωτοβουλίας που βασίζεται στην πράσινη βίβλο της Κομισιόν. Ζωάν Μαρία, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια σε εσά και στου ε, συναδέλφου σα, ε, με του οποίου θα συνεργαστούμε βεβαίω πολύ στενά για αυτή τη δεύτερη θητεία που μα απομένει. Το πιο χαρακτηριστικό φαινόμενο της τελευταίας δεκαετίας είναι βεβαίως ε, ο εμπλουτισμός ε, του ε, οπτικοακουστικού πεδίου στην Ευρώπη με την ανάπτυξη όλων των τεχνολογιών που αφορούν αυτόν τον τομέα και βεβαίως διεύρυνση της προσφοράς οπτικοακουστικού υλικού στους Ευρωπαίους πολίτες με τις νέες προοπτικές και δυνατότητες που τους προσφέρει τόσο στον καταναλωτή όσο και στον ε, δημιουργό. Η πρόσβαση στον πολιτισμό βεβαίως έχει εξελιχθεί ιδιαίτερα με την αλλαγή την, ε, ε, του, του υλικού και την εξέλιξη του διαδικτύου που βεβαίως επιφέρει και πολλές προκλήσεις, έχει δημιουργήσει πολλές προκλήσεις σε αυτόν τον τομέα. Θεωρώ ότι είναι καλό ότι η, νομική η ένομη ε, προσφορά του οπτικοκοστικού υλικού ε, στο διαδίκτυο προοδεύει συνεχώς με πολλές δυνατότητες που προσφέρονται μέσω αυτής της αγοράς του οπτικοκοστικού υλικού στο διαδίκτυο. Με αυτές τις παρατήρησει λοιπόν αποφάσισα και εγώ να επικεντρωθώ πιο συγκεκριμένα στην ε, καθιέρωση συγκεκριμένων στρατηγικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την διευκόλυνση ε, της ε, προσφοράς του κοκκουστικού γλυκού στο διαδίκτυο, κινηματογραφικού βεβαίως, υπογραμμίζοντας τον πολύ σημαντικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ε, καθιέρωση μια πραγματική ευρωπαϊκή αγορά σε αυτό το τομέα και βεβαίως μένουν ακόμα πολλά να γίνουν. Η πρώτη μου διαπίστωση είναι ότι η εξέλιξη του νομικού, ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου που θα ε, ευνοήσει και θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων και την ε, εύκολη πρόσβαση στους Ευρωπαίους πολίτες είναι ένα απαραίτητο στοιχείο θα πρέπει να έχουμε κατά νου την, ε, τον μεγάλο πλούτο και τη μεγάλη κληρονομιά που έχουμε σε οπτικοακουστικό επίπεδο, επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του και την ε, προώθησή του. Εξάλλου έκανα την επιλογή να μην μείνω στα, στα ζητήματα που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα. Σε αυτά θα επικεντρωθεί ο συνάδελφος κ. Μπορής που είναι εισηγητής ε, από την Νομική Επιτροπή. Βεβαίως, ε, αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας των ε, των δικαιωμάτων διανοητική ιδιοκτησία. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε μια ασφάλεια δικαίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε αυτό το τομέα ε, σε ό,τι αφορά την αγορά αυτή στο διαδίκτυο και να αποφύγουμε τη διακριτική μεταχείριση μεταξύ των υπηρεσιών στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου. Είμαι πεπισμένος ότι θα πρέπει να ε, δημιουργήσουμε μια ενιαία αγορά και για το οπτικοακουστικό υλικό και για το κινηματογραφικό υλικό και όλα αυτά να τα συνδυάσουμε μαζί με την σημασία ε, που έχει να σαβαστούμε την ε, ποικιλομορφία και τη διαφορετικότητα θα πρέπει να αναπτύξουμε την οικονομία του πολιτισμού μέσω μιας ε, φιλόδοξης ψηφιοποίησης, γενικευμένης και υπεύθυνη ε, ψηφιοποίησης του οπτικοκουστικού υλικού που αποτελεί τμήμα της κληρονομιάς μας ε, μέσω των της Ευρωπαϊκή της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης και άλλων μέσων και μέτρων που αναλαμβάνονται από τον τομέα του οπτικοκουστικού και κινηματογραφικού υλικού με το ESAN, International Standard Audiovisual Number, αυτό τον ε, ε, διεθνή αριθμό. Για να υπάρχει δηλαδή ένα κάποιο είδους ε, DNA του κάθε έργου. Η επέκταση της ε, αναγνώρισης της χώρας προέλευσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.2 της Οδηγίας ε, ε, του Single Market Act σε σχέση με τις καταχρηστικές ε, μετατοπίσεις θα πρέπει και σε αυτό να δώσουμε σημασία. Μεγαλύτερο ρόλο θα πρέπει να δώσουμε και, στον, ε, και στην παιδεία για να δημιουργήσουμε και μια νέα γενιά που θα σέβεται περισσότερο αυτά τα δικαιώματα. Η παιδεία που αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που βλέπουμε ότι αποφέρει καρπούς τώρα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να χρησιμοποιήσουμε το καλύτερο και πιο ολοκληρωμένο τρόπο ε, τα, το οπτικοκοστικό αυτό υλικό. Είναι επίσης απαραίτητο η πάροχη υπηρεσιών υπηρεσιών εκτός διαδικτύου να προωθούν με τα κατάλληλα μέσα την παραγωγή ευρωπαϊκών έργων μέσω της ε, ε, οικονομικής τους ε, προσφοράς, με την απόκτηση δικαιωμάτων για αυτά τα έργα και με την ύπαρξη τέτοιων έργων στους αντίστοιχους καταλόγους. Η δημιουργία και η ποιότητα θα πρέπει να αναγνωρίζεται πάντα στα πλαίσια αυτής της βιομηχανίας και όλα αυτά απαιτούν μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών και βεβαίως ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορώ να πω ότι δεν θα πρέπει να, να αλλάξουμε αυτό το τομέα με δραστικό τρόπο. Πιστεύω όμως ότι μπορούμε να εξετάσουμε κάποιες τροποποιήσεις. Ε, δηλαδή, να μην χαλάσουμε ό,τι έχει ήδη δημιουργηθεί, απλώς να το προσαρμόσουμε και ε, στα σύγχρονα δεδομένα και στη κατάσταση. Ε, αυτή τη στιγμή εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό δίκαιο ε, και δικαίωμα της ε, αποζημίωσης των κατόχων δικαιωμάτων, ωστόσο δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να επιβάλλουμε μέσω της υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης τέτοια δικαιώματα θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάποια ευελιξία σε αυτό το τομέα. Από την άλλη, και προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτή η ενιαία αγορά θα μπορέσει πράγματι να καθιερωθεί, θα ήταν καλό να μεριμνήσουμε τόσο ώστε οι εταιρείε συλλογική διαχείριση να χρησιμοποιούν ε, ε, συμβατά μεταξύ του μέσα και μάλιστα και τα ίδια. Αυτό θα ήταν το καλύτερο. Τέλο, να σα διασφαλίσω ότι θα επιμείνω στην ανάγκη, στην ανάγκη συνέχισης ενός φιλόδοξου προγράμματος για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, παρά τις διάφορες φήμες που μας έχουν ανησυχήσει και επιμένω στο γεγονός ότι είναι αναγκαίο το πρόγραμμα αυτό για τα μίντια να εξακολουθήσει να υπάρχει με μέσα που θα αφορούν αποκλειστικά και μόνο τον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων. Πιστεύω ότι παρόλο που έχω εργαστεί ε, σκληρά σε αυτό το τομέα, υπάρχουν ακόμα κάποια στοιχεία που θα πρέπει να κάνουμε και βεβαίως θα σας τα παρουσιάσω όταν ε, έρθει η ώρα. Θα είμαι διαθέσιμος βεβαίως ε, πάντα και ο εισηγητής και οι Σκιώδης για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και ευχαριστώ τους συναδέλφους που έχουν ήδη εκφράσει τον ενδιαφέρον τους και μου ε, εξέφρασαν τις απόψεις τους. Τους ευχαριστώ βεβαίως και βεβαίως και θα τα λάβω όλα αυτά υπόψη. Τέλος, ένα εργαστήριο προβλέπεται λογικά και σας ευχαριστώ που το έχετε ε, λάβει υπόψη στις 28 Ιανουαρίου. Και οποια από εσάς θα ήθελαν ε, να έρθουν. Θα σας δώσω ε, περισσότερες ε, πληροφορίες σε μερικές ημέρες. Είμαι και πάλι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και συνάδελφοι. Ευχαριστώ, κύριε Καβαντά. Νομίζω ότι έχετε δημιουργήσει μια πολύ ευρία βάση, μια βάση η οποία έχει και εύρος και βάθος. Νομίζω ότι έχουμε αρκετό υλικό για συζήτηση. Κυρία Τρίπερ πρώτα. Ευχαριστώ Ντόρις, ευχαριστώ κύριε Καβαντά για την ε, παρουσίασή σας. Θα συνεχίσω στα γερμανικά. Αν σκεφτεί κανείς τα θέματα της παρουσίας ε, στο διαδίκτυο των ε, οπτικοακουστικών έργων, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές διαμάχες. Η Mega Upload έκλεισε την προηγούμενη εβδομάδα από την Αμερικάνικη Δικαιοσύνη και μέσα στην συζήτηση για την επανάσταση του διαδικτύου βλέπουμε τις δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους που συμπεριλαμβάνει. Κατά την άποψή μου μπορώ να πω πολύ θετικά πράγματα ότι αυτή η ψηφιακή επανάσταση δίνει τη δυνατότητα σε καλύτερη πρόσβαση σε οπτικοακουστικά έργα, σε έργα τα οποία ήταν μέχρι τώρα προστατευμένα και δεν είχαν καμία δυνατότητα πρόσβασης. Υπάρχει δυνατότητα νέων έργων, υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθούν νέες μορφές δημιουργικότητας και υπάρχουν φυσικά και σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα, νέε εταιρείε, 4 εκατομμύρια θέσει απασχολήσεω που έχουν δημιουργηθεί χάρη σε αυτή τη δραστηριότητα του διαδικτύου. Επομένω, όλα αυτά τα θέματα είναι πολυθετικά και είναι προφανέ ότι ο κόσμο είναι πολύ διαφορετικό τώρα το 2012 από ό,τι ήταν το 1990 με τι δυνατότητε να έχουμε ε, ανταλλαγή και αντιγραφή έργων με τα smartphones, με, τις, με τους ε, υπολογιστές ταμπλέτες, αλλά φυσικά υπάρχουν και δυνατότητες για παράνομες δραστηριότητες και αυτό μας φέρνει στο πρόβλημα αυτό το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Για μένα το σύστημα είναι να κάνουμε μία διάκριση μεταξύ πληροφοριών που μπορεί κανείς να ανταλλάξει επίσημα και για πληροφορίες που έχουν πολιτικό χαρακτήρα φυσικά δεν μπορεί να υπάρχει καμία μορφή λογοκρισίας. Οι Creative Commons έχουν εργαστεί για να μπορεί να υπάρχει αυτή η δυνατότητα αδειών χρησιμοποίησης αυτών των έργων και αυτό συμβάλλει στην ψηφιακή επανάσταση και στην ψηφιακή ανάπτυξη της γνώσης. Τα έργα λοιπόν αυτά τα οποία βρίσκονται στο δημόσιο χώρο, όταν υπάρχει μεταλαμπάδευσή τους, αυτό δεν είναι καθόλου πρόβλημα και αυτό το έχουμε συζητήσει και αποφασίσει στα πλαίσια της συζήτησης έκθεσης Ευρωπαίανα. Όταν όμως υπάρχουν περιεχόμενα τα οποία προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών τους, εδώ τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα. Και εδώ θα πρέπει να βρούμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ απλό με ένα κλικ του ποντικού κανείς να αντιγράψει αυτά τα έργα, να τα αποστείλει, να υπάρξει ιδιωτική ανταλλαγή μεταξύ ατόμων, κάτι πολύ διαφορετικό από την εμπορική χρήση και μεταλαμπάδευση αυτών των έργων. Όλα αυτά λοιπόν απαιτούν μια καλύτερη σκέψη για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να υπάρχει η ανταμοιβή των καλλιτεχνικών δημιουργών. Γιατί μας ενδιαφέρει να υπάρξει και αναγνώριση αυτής της δημιουργικής δραστηριότητας που είναι και η βιοποριστική πηγή για τους καλλιτεχνικούς δημιουργούς, τουλάχιστον για πολλούς από αυτούς, και να υπάρχει δυνατότητα ανταμοιβή για τα έργα τους, όπως γίνεται και με άλλα καταναλωτικά προϊόντα η κοινωνία αποδίδει αξία σε τα θέματα αυτά, επομένως <clears throat> θα πρέπει να υπάρχει και κάποια πληρωμή για τα θέματα αυτά. Είναι πολλά δημόσια αγαθά τα οποία έχουν ελεύθερη πρόσβαση, αλλά εκεί η κοινωνία είναι αυτή η οποία μέσα από τη φορολογία ανταμείβει τους δημιουργούς αυτών των έργων που βρίσκονται στο δημόσιο τομέα. Επομένω, σε ό,τι αφορά τις αγορές πολιτιστικών προϊόντων, είναι απαραίτητο να υπάρξουν νέες νομικές ρυθμίσεις, νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Αυτό το έδειξε ήδη ο τομέα της μουσικής, όπου υπήρξαν και προτάσεις για χρήση αυτών των έργων που δεν ήταν παράνομες. Η Γερμανία έχει ήδη 60 τέτοιες ε, μορφές παρουσίασης έργων οι οποίες είναι σε επίπεδο ε, παράνομο και αυτό δείχνει το πόσο μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχουν για τα θέματα αυτά. Επομένως, είναι απαραίτητο να δώσουμε την πρέπουσα σημασία στα πολιτιστικά έργα, γιατί θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει η σωστή ανταμοιβή, όπως είπα, των καλλιτεχνικών δημιουργών. <clears throat> Υπάρχουν και κάποιοι καλλιτέχνες οι οποίοι κάνουν το έργο τους προσβάσιμο σε όλους, γιατί αυτό είναι και μια μορφή διαφήμισης, αλλά το να γίνεται κάποια χρησιμοποίηση αυτών των έργων σε βάρος τρίτων όπως έγινε από τη Mega Upload, αυτό πιστεύω ότι δεν είναι σωστό. Και λέω και εγώ πάλι ότι δεν αποσκοπώ σε κάποια μορφή πολιτικής λογοκρισίας, δεν θέλω να υπάρξει καμία καταποίηση της πολιτικής ελευθερίας έκφρασης, αλλά με ενδιαφέρει να υπάρξει η προστασία των καλλιτεχνικών δημιουργών και του έργου τους και να υπάρχει η δυνατότητα να εμποδίσουμε τρίτους να αποφελούνται με κλιματικό τρόπο από τα έργα αυτά. Είσαστε Γάλλος και η Γαλλία έχει αντιμετωπίσει ήδη πολλές διαμάχες για τα θέματα αυτά. <clears throat> Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ε, είναι λαθασμένο να στρεφόμαστε κατά του τελικού χρήστη και αυτό φαίνεται και από υποθέσεις που βρίσκονται αυτή στα, δι, δικαστήρια. Καλύτερα να στρεφόμαστε εναντίον αυτών οι οποίοι προσπαθούν να εμπορευθούν αυτά τα καλλιτεχνικά έργα και να τα εκμεταλλευτούν και αυτό θα ήταν πολύ καλύτερο να το κάνουμε και συνοδευόμενο από μια εκστρατεία που θα καταδείξει ότι τα πολιτιστικά αυτά προϊόντα θα πρέπει να έχουν το αντίστοιχο τίμημα και όχι να είναι δωρεάν ή ιονίδιο δωρεάν με τον τρόπο αυτό μπορεί και η ψηφιακή οικονομία να βοηθήσει να βρούμε νέους τρόπους να καταλογίσουμε τίμημα για αυτά τα προϊόντα, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι όλα αυτά τα έργα θα πρέπει να έχουν μία ανταμοιβή με έναν τρόπο ο οποίο πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες ψηφιακές συνθήκες. Μίλησε και για την εσωτερική αγορά ο κ. Καβαδά και τόνισε τη σημασία της εσωτερικής αγοράς και την επέκταση της αγοράς αυτής και στα καλλιτεχνικά προϊόντα και την επιγραμμική μετά ε, διανομή τους. Αλλά από την άλλη δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε ορισμένου τομείς όπω η μουσική υπάρχει μια επικυριαρχία κάποιων εταιριών αγγλοσαξονικών οι οποίες έχουν καταφέρει να επεκταθούν σε όλη την Ευρώπη και να εκτοπίσουν άλλες εταιρείε τοπικές Και αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δεν μου φαίνεται ότι είναι δυνατό να υπάρξει μια πανάκια, μια λύση σε όλους τους τομεί. Δεν θα ήθελα τώρα να μπω στι λεπτομέρειε η μουσική έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα. Απλώς πιστεύω ότι ο τομέας αυτός χρειάζεται περισσότερο εμβάθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Εβετ, Κάμερα Εβετ μάλλον. Σας ευχαριστώ και εγώ. <clears throat> Ευχαριστώ και τον κύριο Καβαντά για την παρουσίασή του. Προφανώς δεν μπορούμε να παρακάμψουμε τα προβλήματα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τα πνευματικά δικαιώματα. Είναι θετικό όμως το γεγονός ότι δεν καλύπτει το σύνολο αυτής της προβληματικής ή προβληματική των πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να αντιμετωπίσουμε και άλλα θέματα τα οποία και αυτά συνδέονται γενικά με τα οπτικοακουστικά μέσα και την χρήση σε επιγραμμικό επίπεδο αυτών των οπτικοακουστικών μέσων. Νομίζω ότι έχουμε κάνει ήδη μια πολύ καλή προπαρασκευαστική εργασία. Αναφέρομαι στην έκθεση του συναδέλφου Μπέλετ για τα συστήματα αυτά, τα οπτικά οπτικοακουστικά και εκεί υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία μας απασχολούν και τώρα τα οποία είχαν ήδη αντιμετωπιστεί πρώιμα. Βρισκόμαστε λοιπόν στην πολιτική σε μια κατάσταση που τρέχουμε τον ε, τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις γιατί η τεχνολογία προχωρά πάντα πολύ πιο γρήγορα από την διαμόρφωση απόψεων. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε να σκεφτούμε και τις ενδιάμεσες, ε, εν, τις ενδεχόμενες μορφές περιορισμού που μπορούν να προκύψουν για τους ραδιοσταθμούς, παραδείγματος χάρη, από την ε, ε, πρόταση της Κομισιόν. Πιστεύω ότι αυτές οι προτάσεις δεν αντιμετωπίζουν ακόμα πλήρως τις ανάγκες του διαδικτύου. Και αυτή τη στιγμή οι δημόσιοι ραδιοσταθμοί βρίσκονται κάτω από πολύ αυστηρότερες προδιαγραφές από ότι οι ιδιωτικοί, οι ελεύθεροι ραδιοσταθμοί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε με δύο οπτικές γωνίες στον οπτικο-ακουστικό τομέα. Προφανώς είναι ένα εμπορικό αγαθό όλα αυτά τα οπτικοακουστικά προϊόντα, αλλά μιλάμε συγχρόνως πάντα για ένα πολιτιστικό αγαθό. Αυτός ο διτός χαρακτήρας λοιπόν θα πρέπει να μας κάνει να καταλάβουμε ότι είναι διαφορετικά από το ψωμί, το γάλα ή τη γαρδούμπα τα πολιτιστικά αγαθά που έχουν μονάχα ένα εμπορικό χαρακτήρα. Και αυτό θα είναι χρήσιμο να το υπογραμμίσουμε σε αυτή την έκθεση. Σε ό,τι αφορά το copyright, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε και πιστεύω ότι πέραν όλων των ε, προσπαθειών να επιτύχουμε μια ισορροπία που ανέφερε η κυρία Τρίπελ, είναι απαραίτητο να βρούμε πώ θα μπορούμε να έχουμε και ένα σύστημα το οποίο είναι εύληπτο και απλό και το οποίο να μπορέσει να λειτουργήσει σε όλη την Ευρώπη και να οδηγήσει σε σαφήνεια δικαίου. Και επίσης υπάρχει και η ανάγκη μιας παιδαγωγίας σε σχέση με τα μέσα ενημέρωση. Πώς μπορούμε να, να πείσουμε τους πολίτες ότι τα πολιτιστικά αγαθά έχουν μία αξία και πρέπει να καταβάλουν το τίμημά τους. Όχι μόνο λοιπόν να έχουμε μια κατασταλτική ε, και κολαστική ε, αντιμετώπιση, αλλά να εξηγήσουμε και την αξία του. Κάτι άλλο το οποίο μου φαίνεται σημαντικό είναι το θέμα της φορολογίας. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να επηρεάσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και εδώ νομίζω ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι είναι παράλογο τουλάχιστον στη Γερμανία ότι η εφημερίδα που αγοράζει κανείς στο περίπτερο πληρώνει 7% ΦΠΑ αλλά σε, σε μία ε, άλλη μορφή πώληση εφημερίδας μέσω επιγραμμικών συστημάτων μπορεί να είναι 19% το ΦΠΑ, αλλά δεν υπάρχει καμιά ουσιαστική διαφορά. Γιατί το ένα σύστημα να υπόκειται σε υψηλότερο ΦΠΑ. Είναι λοιπόν απαραίτητο να προχωρήσουμε και σε αυτά τα εφή μοντέλα, μοντέλα τιμολόγησης που ανέφερε η κυρία Τρίπερ και τα οποία να περιλαμβάνουν και μια ισοδίκαια φορολόγηση. Είναι ένα από τα παραδείγματα λοιπόν πραγματών που θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για αυτά. Ελπίζω λοιπόν ότι μέσα από την παρουσίαση του κυρίου Καβαντά την πρότασή του και με τις συζητήσεις στην Επιτροπή μας θα μπορέσουμε εν καιρό να καταλήξουμε σε μια πλήρη και συνεκτική έκθεση και ελπίζω ότι αυτή θα είναι και η πραγματικότητα. Ευχαριστώ. κύριος Λόκεγκάρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχηθώ καλή χρονιά στους συναδέλφους. Πράγματι, το θέμα αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Καβαδά, για την τόσο καλή παρουσίαση του θέματος. το θέμα αυτό περιέχει δύο από τα πλέον αγαπημένα ε, μου θέματα που είναι και η πολιτιστική διάσταση της Ευρώπης και η εσωτερική αγορά από την άλλη και ελπίζω πραγματικά το θέμα αυτό να τύχει μια ισορροπημένη αντιμετώπιση. Πολλά ήδη είπαν ε, οι συναδελφοί μου και οι ηγητές. Ήθελα και εγώ να προσθέσω με τη σειρά μου λίγα λόγια ακόμη και να πω πρώτα απ' όλα όταν μιλάμε για διασυνοριακή μετάδοση ραδιοφωνικών και τροπτικών σταθμών, σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε το κατάλληλο περιβάλλον ώστε να μπορεί να γίνει διασυνοριακά αυτό και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να ικανοποιούμε τα αιτήματα των καταναλωτών σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Όχι μόνο για να ενισχύσουμε όσο γίνεται περισσότερο το δυναμικό της ενίας αγοράς, αλλά και για να μπορέσουμε να δώσουμε και μεγαλύτερη έμφαση στην ε, πολιτισμική ποικιλομορφία που είναι και ένας από τους στόχους της Επιτροπής μας. Δεύτερο, κατακαιρματισμός. Ε, πρέπει να βρούμε λύσεις για να αντιμετωπίσουμε τον κατακαιρματισμό των επιγραμμικών αγορών, ιδίω. Αναφέρουμε στο θέμα της αδειοδότησης ε, που γίνεται επιγραμμικά, είναι κάτι που έθεσαν και άλλοι συνάδελφοι. Ξέρετε, σε έναν ιδανικό κόσμο δεν θα έπρεπε να έχουμε να αντιμετωπίζουμε 27 διαφορετικά καθεστώτα. Και αυτό, ξέρετε, ο κατακαιρματισμός οδηγεί σε μη σαφείς κανόνες για την αντιμετώπιση και προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν καλές προτάσεις. Ε, ήδη υπάρχει μια μακρά και σκληρή εργασία είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει και τη δική μας Επιτροπή για να μπορέσουμε να βρούμε τι κατάλληλε λύσει. Τρίτον, κάτι που ήδη υπόθηκε και πάλι, είναι το θέμα των αμοιβών. Δηλαδή, οι δημιουργοί θα πρέπει να αμείβονται ικανοποιητικά ώστε να μπορούν να ασκούν και βιοποριστικά, αν θέλετε, την τέχνη τους και να πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο με απασχολεί εδώ και καιρό και παρακολουθώ α, τις εξελίξεις ε, για μεγάλο διάστημα. Είναι πραγματικά σύνθετο το ζήτημα και ναι μεν ε, η διαδικασία ω τώρα ήταν δύσκολη και σύνθετη, όμως πιστεύω ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά και προσβλέπω σε μια καλή συνεργασία με τον εισηγητή και τους ε, ε Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον κύριο Καβαντά για το έργο το οποίο έχει φέρει σε πέρας. Πιστεύω ότι οι προτάσεις που έχει παρουσιάσει σήμερα μέσω της έκθεσής του πηγαίνουν στη σωστή κατεύθυνση. Το θέμα του copyright δεν μπορούμε βέβαια να το αποσυνδέσουμε από το σύνολο της προβληματικής για τα θέματα αυτά, αλλά θα πρέπει συγχρόνως να κάνουμε σαφές ότι οι κανόνες οι οποίοι για μας είναι φυσιολογικοί στον μη επιγραμμικό τομέα θα πρέπει να ισχύουν και στον τομέα του, τον επιγραμμικό. Δηλαδή να έχει κάνει το δικαίωμα να κάνει μια, ένα αντίγραφο μονάχα για προσωπική χρήση. Αλλά βέβαια δεν είναι το ίδιο πράγμα το ίντερνετ όπως το να κυκλοφορεί κανείς με ένα με μια μηχανή βίντεο και να φιλμάρει την, ε, το γύρο του και με τον τρόπο αυτό να μπορεί να παίρνει πληροφορίε. Λοιπόν, πρέπει να υπάρξει αυτή η προστασία στο ίντερνετ, είτε είναι κάτι εμπορικού χαρακτήρα, είτε μη εμπορικού χαρακτήρα. Υπάρχει μια τεράστια, μια τεράστια δραστηριότητα ανταλλαγή και αντιγραφή ε, ταινιών που δεν θεωρούνται πια σχεδόν να είναι ιδιωτικά προϊόντα, να είναι καλλιτεχνικά προϊόντα. Επομένως αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το επιλύσουμε από τη μια μέρα στην άλλη. Θα πρέπει να ουσιαστικά να αποδεχθούμε ότι έχουμε αφήσει αυτό το τομέα να είναι ένας χώρος αναρχίας χωρίς καμία απολύτως ε, ρύθμιση. Οι νέοι έχουν συνηθίσει μια τέτοια κατάσταση και θα πρέπει να τους πείσουμε να έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση. Η αύξηση των ε, επιγραμμικών προϊόντων έχει οδηγήσει σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα, έχει αλλάξει και τους τρόπους με τον οποίο γίνεται η καταβολή κάποιου αντιτίμου. Θα πρέπει να έχουμε μια νέα συνείδηση για τα προϊόντα αυτά, ώστε ο χρήστης αυτών των προϊόντων στο διαδίκτυο και η γενιά αυτή η οποία έχει μεγαλώσει με τους υπολογιστές να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο το βλέπει αυτά τα προϊόντα. Είναι απαραίτητο λοιπόν όλα αυτά να γίνονται με έναν τρόπο ο οποίος είναι σαφής και ισορροπημένος και πιστεύω ότι αυτά τα οποία είπε και παρουσίασε ο Ζωάν Μαρικαβαντά. Είναι μια σειρά από θετικές προτάσεις που μπορούν να δώσουν ε, σάρκα και οστά σε μια ευρύτερη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η συζήτηση θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Τα πιο πολλά που ήθελα να πω ήδη τα είπαν οι προλαλήσαντες και έθεσαν πολύ καλά τη βάση της συζήτησης. Θα ήθελα μόνο εγώ από πλευρά μου να θέσω ένα απλό θα έλεγα ζήτημα που μπορεί να είναι, αν θέλετε, η επόμενη κρίση σχετικά με την επιδημική διανομή περιεχομένου. Συνήθω προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την τελευταία κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει, δηλαδή την κρίση στην πρόσβαση που αφορά την υπερβολική δυνατότητα πρόσβαση αν θέλετε, σε τέτοιο υλικό, που αφορά μεμονωμένους καταναλωτές που έχουν υπερβολική πρόσβαση σε αυτό το οπτικοακουστικό ε, υλικό. Μπορεί όμως η επόμενη κρίση να είναι πολύ διαφορετική, να είναι πολύ πιο συγκεντρωτική και να αφορά πιο πολύ την πλευρά των διανομέων. Τουλάχιστον βιομηχανίες, για παράδειγμα. Να δώσω να πω κάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα η Apple παρουσίασε τρία εργαλεία που από ό,τι κατανοώ το επόμενο διάστημα θα δώσουν νέους όρους στη συζήτηση, για παράδειγμα. Τα νέα σχολικά βιβλία που θα μεταδίδονται μέσω των tablets και των iPhones. Περίεργο φαίνεται, γιατί αυτό το σχολικό βιβλίο θα περιέχει οπτικοακουστικό ε, υλικό και θα περιέχει μουσικά στοιχεία, διαδραστικά στοιχεία, ε, φιλμ κτλ. Και έχει κάτι άλλο επίσης πολύ ενδιαφέρον. εγώ θεωρώ ότι είναι εξαιρετική η ιδέα που μας είπε ο κ. Πεβατάνη προκειμένου, ότι έχει τη δυνατότητα να επικαιροποιείται συνεχώς. Δηλαδή, εγώ δημοσιεύω ένα βιβλίο και θα πρέπει να ε, έχω συνεχώς νέες εκδόσεις για να το ενημερώνω. Ενώ με αυτό το βιβλίο το επιγραμμικό θα επικαιροποιείται ε, με το πάτημα ενός κουμπιού. Και αυτόματα όλοι θα λαμβάνουν αυτή την ενημέρωση. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν θα υπάρχει συνεχώς επικαιροποίηση μέσω του λογισμικού αυτών των βιβλίων. Δεύτερο στοιχείο που θέλω να αναφέρω, νέο εργαλείο της Apple, είναι ένα εργαλείο για την αυτοδημοσιευση ένα self-publishing. Δηλαδή, ο δημιουργός ολοκληρώνει το έργο, το βιβλίο του, ε, στο οποίο μπορεί να εντάξει τα γραφικά στοιχεία, τα φίλου και οτιδήποτε άλλο έχει ως οπτικοστικό υλικό. Πατάει ένα κουμπί, λέει publish για δημοσίευση και μέσω της Apple ε, θα ε, γίνει δημοσίευση και έπειτα τα κέρδη θα πηγαίνουν 50% για παράδειγμα στην Apple και το 50% σε αυτόν. Τι θα σήμαινε κάτι τέτοιο αυτό και πώς σχετίζεται με το θέμα που συζητούμε. Ναι, η κρίση που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια μα έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα. Τι μπορεί να μα συμβεί στο μέλλον. Τέτοια εργαλεία τη Apple φυσικά θα χρησιμοποιηθούν και μέσω τη Amazon. Όμω, ξέρουμε ότι πολύ συχνά αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιούνται καθαρά εν είδη μονοπωλίου. Φοβούμε ότι μονοπωλιακά τέτοιου είδους εργαλεία self-publishing θα χρησιμοποιηθούν το πολύ. Ένας ή δύο δηλαδή θα έχουν το μονοπόλιο για τη χρήση ε, επιγραμμικά αυτών των νέων εργαλείων. Και Ξέρετε, βέβαια, αυτό το εργαλείο μπορεί να είναι εξαιρετικό και φυσικά πάρα πολλοί δημιουργοί θα χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο για να δημοσιεύσουν επιγραμμικά τα βιβλία τους και να μπορούν να λαμβάνουν, αν θέλετε, ε, πολύ πιο άμεσα τα κέρδη και τις αμοιβέ από την πώληση των έργων αυτών. Όμως αυτό ε, θέτει ένα αμφιβόλο και τον τρόπο τον οποίο θα ενημερώνονται και θα τροποποιούνται και οι συμβάσεις που θα έχουν οι δημιουργοί και αυτό το ισχύει και ως πρόβλημα και για τα επιστημονικά περιοδικά. Δεν προσπαθώ να εξάγω κάποια συμπεράσματα, απλά θέλω να θέσω κάποια α, στοιχεία ως τροφή για σκέψη και συζήτηση. Και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα νέο κύμα υπηρεσιών που θα δημιουργήσει και μια νέα κρίση. Θέλω να πω δηλαδή ότι ενώ τώρα είχαμε τον κατακαιρματισμό, στο μέλλον μπορεί να έχουμε πιο πολύ πρόβλημα μονοπωλιακό. Και τέλος, για να μπορούμε να εντοπίσουμε καλύτερα αυτά τα βιβλία, να ταυτοποιούμε καλύτερα αυτά τα βιβλία, χρειαζόμαστε, πιστεύω, μια καλύτερη μορφή του ESSEN για να μπορούμε να ταυτοποιούμε καλύτερα αυτά τα έργα. Εξαιρετική λοιπόν η ιδέα του ESIN, e γιατί είναι μια, ένα απλό εργαλείο και πιστεύω ότι θα είναι πολύ χρησιμοποιημένο και τις βιβλιοθήκες του μέλλοντος. Ευχαριστούμε κύριε Ταβάρες, πολύ ενδιαφέροντα τα λεγόμενά σας. Κυρία Μακλάφλιν. Κλάκλιν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Καβαντά για την παρουσίασή του, για την επιγραμμική διανομή των κακοστικών έργων. Όλοι εδώ πέρα σε αυτή την Επιτροπή γνωρίζουμε πόσο ε, σημαντική είναι αυτή η βιομηχανία, δισεκατομμύρια ε, εσόδων, αλλά και εκατομμύρια, εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Υπάρχει όμως και πραγματική ζήτηση από τους πολίτες μας. Εμείς πρέπει όμως να διασφαλίσουμε ότι ότι αξιοποιούμε στο έπακρον αυτό το μέσο, αλλά μεριμνούμε και για την υπεράσπιση των ε, πνευματικών δικαιωμάτων. Πολλές επιπλοκές υπάρχουν όταν έχουμε αδειοδότηση για το copyright. Και για αυτό το copyright ε, ε, για τους συγγραφείς είναι ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία. Σε αυτό το νέο πλαίσιο λοιπόν θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό το ζήτημα, πώς θα μειώσουμε το διοικητικό άκτος και το κόστος όμως. Για να μειώσουμε τον αριθμό όσων ε, ε, κατεβάζουν εντό εισαγωγικών παράνομα οπτικοπιστικό υλικό. Αυτό το σύστημα που ανέφερε ο κ. Καβαντά ε, ενδεχομένω να παράσχει, να παράσχει λύσεις, αλλά μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα. Βεβαίως όμως και ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σα, κύριε Καβαντά και με του υπόλοιπους κοιόδη ε, εισηγητές. Ευχαριστώ. Thank you. Ε, Madam Sanchez Smith. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον συναδελφό μου τον Σαν Μαρή Καβαντά, ο οποίος νομίζω ότι έχει διεξέλθει όλα τα βασικά στοιχεία της προβληματικής αυτής. Είναι πράγματι πολλής χρόνος που διέρευσε χωρίς να εφαρμόσουμε κάποια κανονιστική, κάποιο κανονιστικό πλαίσιο στην επιγραμμική διανομή οπτικο-ακουστικών έργων και ως αποτέλεσμα βρισκόμαστε σήμερα σε μια κατάσταση η οποία δεν απλή. Είναι δύσκολα τα προβλήματα αυτά. Το να έχουμε κάποιο πλαίσιο κανονιστικό στο ψηφιακό χώρο εμπλέκει την πολιτική, την νομική αλλά και την τεχνική πτυχή. Μιλήσαμε για προστασία δικαιωμάτων, για αδειοδοτήσεις συνολικού χαρακτήρα, συλλογικού χαρακτήρα ή εδαφικού χαρακτήρα τουλάχιστον, το να υπάρξει σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων αλλά και μεταλαμπάδευση των έργων αυτών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια πανάκια που θα επιλύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Θα πρέπει πράγματι, εγώ συμφωνώ με αυτά που ελέτησα, να υπάρξει ένας εκπαιδευτικός και παιδαγωγικός ρόλος για να καταλάβουν οι καταναλωτές ποια είναι τα προβλήματα και επίσης θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια εναντί των νέων και των παιδιών ακόμα που είναι οι μελλοντικοί καταναλωτέ. Ευχαριστώ. Κάποιο από την Κομισιόν θα ήθελε να λάβει το λόγο. Ο κύριο Ζολή. Ευχαριστώ, Helen Όλβεν ονομάζομαι από την ε, Ενότητα Πνευματικών Δικαιωμάτων από την Γενική Διεύθυνση αγορά. Εργαστήκαμε και επί τη Πράσινη Βίβλου που δημοσιεύθηκε σε συμφωνία με τις Γενικές Διευθύνσεις ΕΑΚ και Κοινωνία της Πληροφόρησης. 18 ε, Νοεμβρίου το εκδώσαμε. Είχαμε περίπου 200 απαντήσεις από πολλούς ε, φορείς, είτε δημόσιους, ε, είτε από πολίτες και κάποιους από τους ε, φορείς που συμμετέχουν σε αυτό το τομέα, διανομής, πάροχοι, εκπρόσωποι της βιομηχανίας κτλ. Και αυτή τη στιγμή εξετάζουμε όλες αυτές τις απαντήσεις. Σε αυτό το ερωτηματολόγιο των 27 ερωτήσεων, φανταστείτε 200 απαντήσεις για 27 ερωτήματα. Αυτό παίρνει χρόνο βεβαίως και μέχρι τα μέσα του χρόνου θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα. Όπως ανακοινώσαμε και στην ε, ανακοίνωση του ε, ηλεκτρονικού εμπορίου στις αρχές του μήνα, θα λάβουμε υπόψη και, τα, και την υπόθεση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που ε, είχαμε πέρυσι και με αυτό βάσει αυτά τα συμπεράσματα θα δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Δεν μπορώ να πω πολλά παραπάνω. Με τα χαρά θα θέλαμε να λάβουμε αντίγραφο της ε, ε έκθεσης του κυρίου Καβαδά και θα ακούσουμε τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Πολιτισμού και θα τις ε, λάβουμε υπόψη κατά την ε, κατάρτιση της έκθεσής μας. Ευχαριστώ. Θα σας ρωτήσω κάτι, παρακαλώ. για τα ερωτήματα του κυρίου Ταβάρης. Το θέμα της αυτοδημοσίευσης, το self-publishing λοιπόν. Δεν ξέρω αν έχετε να θέσετε μία απάντηση σε τα θέματα αυτά. Um, Αυτό το ερώτημα δεν έχει ανακύψει. Εφόσον εστιάσαμε περισσότερο την προσοχή μα ε, στον οπτικοακουστικό τομέα. Υπήρξαν ορισμένε παρατηρήσει ε, για τον ε, μουσικό τομέα, αλλά ελάχιστε απαντήσει αφορούσαν τον τομέα της, των εκδόσεων. Ίσως έχετε θέσει στον εαυτό σας ε, λαθασμένες ερωτήσεις ή σας διέφυγε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για σας ακόμα. Και έχετε ακούσει κάποιες παρατηρήσεις σήμερα οι οποίες ίσως δεν περιλαμβάνονται στο δικό σας έγγραφο, ίσως θα πρέπει να τις αξιολογήσετε και βλέπετε ότι υπάρχει πολύ υλικό για την περαιτέρω συζήτηση. Κύριε Φερχάινεν, και εγώ θα ήθελα να θέσω ένα σύντομο ερώτημα ακριβώ για αυτό το θέμα. <clears throat> Από ό,τι κατανόησα, όταν εγώ θέλω να ε, κάνω μια αυτοδημοσίευση, μπορώ να το κάνω με τη συνεργασία της ε, Apple και με το λογισμικό iTunes, αλλά αυτό μπορώ να το κάνω μονάχα με το υλικό της ε, Apple. Γιατί άμα θέλω να τυπώσω ένα βιβλίο, εγώ μπορώ το βιβλίο να το δώσω οπουδήποτε να το τυπώσουν. Κρατάει φυσικά ο εκδοτικό ήχο τα δικαιώματα, αλλά δεν με περιορίζει κάποιο να χρησιμοποιήσω ένα σύστημα ή ένα λογισμικό. Δηλαδή, δεν υπάρχει δομή μονοπωλιακή. Θα πρέπει να προσέξουμε στην περίπτωση της ηλεκτρονικής αυτοδιαφήμισης ότι δεν δημιουργούνται μέσω της Apple, μέσω της Google συστήματα μονοπωλιακά τα οποία θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε δυσκολίες και στο μέλλον. Που συστήματα λοιπόν τέτοια μονοπωλιακά που δεν θα επιτρέψουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό μόνο μέσα στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο θα δημιουργήσουν προβλήματα όταν είναι χρήματα τα οποία παίζονται, όταν παίζονται επιχειρηματικά συμφέροντα, τέτοια προβλήματα πάντα μπορούν να προκύψουν. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ενδιαφέρον και πρέπει και η Κομισιό να εξετάσει το θέμα αυτό. Αλλά σας υπενθυμίζω, είχαμε μία ακρόαση για τα θέματα αυτά είχαμε πει ότι είναι καλό να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να βρει ένα εκδότη θα πρέπει να έχει μια δυνατότητα να δημοσιεύσει μόνος του ένα έγγραφο. Το ίδιο πράγμα με ένα σκηνοθέτη ο οποίος δεν βρίσκει κάποιον παραγωγό για να κάνει, για να παραγάγει ένα φιλμ που βρίσκει κάποιο άλλο τρόπο να το παρουσιάσει αυτό. Καταλαβαίνω ότι όλα αυτά είναι και ο τετραγωνισμός του κύκλου. Αυτά τα οποία είναι καλά για τον τομέα της λογοτεχνίας μπορεί να μην είναι καλά για την ε, για το σινεμά, ό,τι είναι καλό για το σινεμά δεν είναι καλό για τα ντοκιμαντέρ. Δεν είναι πολύ εύκολα αυτά τα πράγματα. Εσείς ίσως μπορείτε με νυφαλιότητα να τα αντιμετωπίσετε καλύτερα. Δίνω και πάλι το λόγο στον κύριο Καβαντά. Αν θέλετε. Δεν θέλετε. Ευχαριστώ, αλλά σε αυτό το στάδιο πράγματι απλώς καταγράφω τις παρατηρήσεις. Okay. Ευχαριστούμε και πάλι κύριε Καβαδά. Ήταν πάρα πολύ διαφωτιστικά όλα αυτά τα θέματα. Ξέρετε ότι έχουμε ένα πρόβλημα με αυτή την έκθεση πρωτοβουλίες γιατί η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων διαμφισβήτησε το θέμα αυτό αλλά φυσικά δεν είναι θέμα μονάχα copyright, είναι ένα πολύ ευρύτερο θέμα. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να επιβάλλουμε την απόψή μας στο σημείο αυτό, κύριε Καβάντα. Σημείο 5 είναι η απαλλαγή 2010 Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίνω το λόγο στον κύριο Λόκεγκαρτ. Κάνουμε το 2012 λοιπόν την απαλλαγή του 2010, κύριε Λόκεγκαρτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λίγα λόγια μόνο. Ελπίζω να έχετε λάβει και να έχετε διαβάσει το κείμενό μου. Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας πάντοτε είναι να ελέγχουμε κατά πόσον ε, ο ευρωπαϊκός προπολογισμός την χάνει της κατάλληλης διαχείρισης. Πριν την απαλλαγή γίνεται μια εντελεχής εξέταση των λογαριασμών. Ε, διαβάσει με μεγάλη προσοχή τη σχετική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και τις ε, απαντήσεις που δίνουν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί και έπειτα ε, ψηφίζουμε, μάλλον εγκρίνουμε ένα σχετικό ψήφισμα. Αυτό που έχετε μπροστά σε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης βασίζεται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου για την εφαρμογή, την εκτέλεση μάλλον του Γενικού Προπολογισμού του Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2010. Επίσης, εξετάσαμε και την έκθεση αιτήσεις δραστηριότητας της ΓΔ Παιδείας Πολιτισμού και τις σχετικές εκθέσεις των εκτελεστικών οργανισμών εκπαίδευσης, οπτικοστικών θεμάτων και πολιτισμού και του οργανισμού που ασχολούνται με τη δράση Marie Curie. Τα πορίσματά μας, κατά κύριο λόγο θετικά, η περισσότερη απλοποίηση και πιο ευέλικτες διαδικασίες, ειδικά αν δείτε τι συμβαίνει στην γάμα δέλτα για θέματα παιδείας. Βλέπουμε ότι το περιθώριο λάθους, σφάλματος, συγγνώμη, είναι κάτω 2% και ο χρόνος χρηματοδότησης είναι πολύ σημαντικό ειδικά για τους δικαιούχους. Κάτι που πρέπει να επισημάνουμε αφορά την διαχείριση της διαβίου μάθησης. Οι σχετικοί φάκελοι θα πρέπει να την χάνουν καλύτερες διαχείρισεις, ώστε να ε, επιλύονται τα σχετικά προβλήματα κάποιων δικαιούχων ταχύτερα θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στου ευρωπαϊκού και στου εθνικού οργανισμού για την εξέβρεση έγκαιρων λύσεων. Σε σχέση τώρα με την καμάλτη επικοινωνία, η όλη έκθεση δεν εντοπίζει προβλήματα για την εκτέλεση του προπολογισμού. Ένα μόνο σχόλιο έχω να κάνω και αφορά το ε, πανευρωπαϊκό τηλεοπτικό δίκτυο. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, απλά θα ήθελα να επισημάνω ότι χωρίς τη συνένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ε, διεκόπη το σχετικό σχέδιο και αποφάσισε η Επιτροπή να διοχετεύσει τα χρήματα αλλού. Αυτά είχα να πω για την απαλλαγή, Πρόεδρε. Σχόλια, παρακαλώ. not to be the case. Thank you very much, Mr. Όχι, οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Λόκεν. Α, με συγχωρείτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Uh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω και να συμφωνήσω την πλειοψηφία των λεγόμενων ε, του εισηγητή, ιδίω ό,τι αφορά τα θέματα επικοινωνία και πολιτισμού. Πραγματικά, κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια στον τομέα απλοποίηση, βελτιώνοντα συστήματα ελέγχου και το ελεγκτικό συνέδριο αναγνωρίζει τον πιο αποτελεσματικό τους πλέον χαρακτήρα. Στο θέμα τη χρηματοδότηση και των πληρωμών πιστεύω ότι επιτυγχάνουμε σημαντική βελτίωση ήδη. Αυτό που επισημαίνει το Λυκό Συνέδριο, ότι υπάρχει ένα τομέα που καλό είναι να υπάρξει μεγαλύτερη πρόοδο. Αυτό αφορά το, τον έλεγχο σε πρώτη φάση για τη διαβίου μάθηση. Πράγματι, συμφωνούμε με αυτό. Να πούμε ότι οι εθνικοί οργανισμοί σε κάποιου τομείς ε, προβαίνουν σε υπερβολικούς ελέγχους. Οπότε συζητούμε με τους εθνικούς οργανισμούς, προσπαθώντας να του πείσουμε ότι ε, δεν πρέπει να υπερβάλλουν στους ελέγχους και θα πρέπει να παραμένουν σε αυτούς που είναι αναγκαίοι. Ε, υπάρχει μια γενική συμφωνία, αλλά πρέπει να υπάρξει και περαιτέρω πρόοδο στον τομέα. Ένα ακόμη τεχνικό σχόλιο σε ό,τι αφορά το κείμενό σας. και τα σχόλια του εισηγητή σας. Λέτε ότι χαιρετίζει το γεγονός, ε, μάλλον διαπιστώνεται με ικανοποίηση ότι δεν έχουν υπάρξει ουσιώδη σφάλματα στο τομέα πολιτικής πολιτισμού και ε, παιδείας. Πράγματι, στατιστικό επίπεδο, ναι, ε, δεν έχουν εντοπιστεί ουσιώδη σφάλματα, δεν έχουν υπάρξει δηλαδή σφάλματα πάνω από 2% για το σύνολο. Δηλαδή, ε, μιλάμε για δραστηριότητες που καλύπτουν και την έρευνα. Αν δείτε τους σχετικούς πινακές, δεν εντοπίσετε ε, ουδένα σφάλμα. Ε, Mr. Nautz, ε, Κύριος Νάουτς, θα ήθελε να πει κάτι όμως για το σημείο 5. To point five of the remarks of Mr. Για το σημείο 5, παρακαλώ, θέλετε. Ευχαριστώ. Ανταγαντζέ, από τη Γενική Διεύθυνση Αρμόδια. Αρχικά θα ήθελα να σας συγχαρούμε για την πολύ ε, θετική στάση του εισηγητή, για την ε, διαχείριση του προϋπολογισμού του 2010. Σε ό,τι αφορά πιο συγκεκριμένα το σημείο 5, συμφωνούμε ή μάλλον έχουμε πλήρη επίγνωση ε, της παρατήρησης του εισηγητή. Ο Γενικός μας ε, Διευθυντής, ε, κύριος Πολζέ, είχε την προηγούμενη εβδομάδα τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει στον εισηγητή ότι θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο σε αυτό το σημείο και θα μεταβιβάσει το σημαντικό δυνατό το σύνολο των ε, εγγράφων που ζήτησε ο εισηγητή για αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λόκογκάρτ. Yes, thank you. Ευχαριστώ. Μία παρατήρηση μόνο σε αυτό που είπατε. Το σημειώνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα ερώτημα έχω για τους ελέγχους που αναφέρατε προηγουμένως. Είπατε ότι είναι πάρα πολύ. Όμως, πώς μπορεί κάποιος από τον προτέρων να γνωρίζει τι είναι έλεγχος και τι όχι. Εμείς ζητήσαμε από τις εθνικές υπηρεσίες να κάνουν ε, ανακατηγορία, αναμορφή ε, δράσης ένα, ένα ελάχιστο αριθμό ελέγχων πριν από την ε, δραστηριότητα, μετά κτλ. Έχουμε θέσει λοιπόν κάποιους όρους και παρατηρήσαμε ότι σε κάποιες εθνικές υπηρεσίες πάνε πέρα από τα όσα ζητούμε ε, σε κάποιους ε, τομείς ελέγχου θέλουν να τα, να τα ελέγξουν όλα. Ενώ εμεί του λέμε δεν χρειάζεται να τα κάνετε όλα, μπορείτε να κάνετε και τα μισά, για παράδειγμα. Ενώ σε άλλου τομεί παρατηρήσαμε ότι δεν φτάνουν στον ελάχιστο αριθμό ελέγχων. Αυτό που εμείς έχουμε ορίσει ως ελάχιστο αριθμό για να έχουμε επαρκή βεβαιότητα. Γιατί αυτό ποικίλει και από, την, από τον τύπο δραστηριότητας, γιατί εξαρτάται και από τον κίνδυνο που εμπεριέχει η κάθε δραστηριότητα. Αν κατάλαβα καλά λοιπόν, δεν πρόκειται για ε, κακή θέληση, απλώς είναι τεχνικό το ζήτημα, πρακτικό. Όχι βεβαίως και δεν πρόκειται για κακή βούληση, μάλλον δεν ε, νιώθουν ήρεμοι να μειώσουν τα επίπεδα ελέγχου τους. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ κύριε Λότεργαρτ κύριε Βόχανζε. Βόχιγκερ στα γερμανικά. Καταληκτική προθεσμία 31 Ιανουαρίου. Για τις τροπολογίες βεβαίως, ε, πολύ σύντομα. Εντάξει, επόμενο σημείο για τις ε, μακροπεριφερειακές στρατηγικές. Κυρία Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θέλω να εκμεταλλευτώ αυτά που είπε ο κύριος Κεγκογκάρτ για να σας ε, συγχαρώ όλους για την εκλογή σας και να σας ευχηθώ τα καλύτερα για τον νέο χρόνο. Έχω αναλάβει λοιπόν τη σύνταξη αυτής της γνωμοδότησης γιατί η μακροπεριφερειακή στρατηγική που έχει ξεκινήσει με απόφαση της Κομισιόν δίνει μια νέα διάσταση στα αποκεντρωμένα περιφερειακά σχέδια συνεργασίας. Και μου φαίνεται ότι κυρία Μπεναράμπ λίγο πιο αργά. Ναι, ναι, έχετε δίκιο, είχαν και διερμηνεί στην αίθουσα. Θα τα πω πιο σιγά. Ο στόχος των μακροπεριφερειών είναι να αρθρώσουν καλύτερους δεσμούς μεταξύ των διαφόρων εδαφικών περιοχών ώστε να εργαστούν καλύτερα και πιο αρμονικά για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν να αντιμετωπίσουν. Αυτή η στρατηγική έχει ήδη αποδείξει την αξία της το 2009 στην περιοχή της Βαλτικής και στην περιοχή του Δουνάβεως το 2010 γιατί ενίσχυσαν την συνεργασία μεταξύ διαφόρων περιφερειών για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν στόχοι οικονομικοί και οικολογικοί. Είναι λοιπόν ένα γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να καθοριστούν προτεραιότητες προγραμμάτων και να κατευθυνθούν οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Θα ήταν πολύ χρήσιμο λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης <clears throat> αυτών των μακροπεριφερειών σε άλλες δραστηριότητες και επίσης και σε άλλες περιοχές οι οποίες και αυτές έχουν μεγάλη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης. Η μακροπεριφερειακή λοιπόν στρατηγική μας φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα εύστοχη για την περιοχή της Μεσογείου. Είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε έμφαση σε αυτήν την ε, περιοχή που είναι το λίκνο της ζωής και του πολιτισμού, όπου και τα γεγονότα της προηγούμενης άνοιξης θα πρέπει να μας ενθαρρύνουν να αναπτύξουμε νέες πιο ενεργές πολιτικές γειτονίες. Παρά τις κοινέ προκλήσεις λοιπόν που βλέπουμε, βλέπουμε να υπάρχει πολύ περιορισμένη συνεργασία και διασύνθεση μεταξύ των περιοχών αυτών. Εξακολουθεί ο κατακαιρματισμός, διαφορετικές πολιτικές καταυθύνσεις που θα πρέπει να ξεπεραστούν με μια κοινή αντιμετώπιση και πολιτική κατεύθυνση. Το μήνυμα αυτό λοιπόν πρέπει να είναι στεναρό, γιατί η θέλησή μας θα πρέπει να είναι η μεταλαμβάδευση γνώσεων και ιδεών, η ενίσχυση της συνεργασίας στον πνευματικό τομέα, και η καλύτερη αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών της Μεσογείου. <clears throat> Είναι απαραίτητο λοιπόν να αντιμετωπίσουμε και τις ε, τάσεις προς μία απομόνωση και μία εσωστρεφή αντιμετώπιση που εμφανίζονται και στις δύο όχθες της Μεσογείου. Μέσα στην γνωμοδότησή μου προτείνω να υπάρξει μια προσέγγιση η οποία θα οδηγήσει σε καλύτερο συντονισμό των ενεργειών της κοινωνίας των πολιτών για καλύτερη προσέγγιση στα πολιτικά αυτά προβλήματα. Δεύτερον, τονίζω την ανάγκη να αυξηθούν οι πολιτιστικές και εκπαιδευτικές ανταλλαγές και οι χώρες της νότιας όχθης Μεσογείου να μπορούν να εποφελθούν από τα κοινοτικά προγράμματα στον τομέα αυτό. Τρίτον, είναι απαραίτητο να υπάρξει μεγαλύτερη κινητικότητα φοιτητών και διδασκόντων και να υπάρξει καλύτερη διαδικτύωση των πανεπιστημίων στην ε, ε, Μεσόγειο χωρίς να δώσουμε μόνο έμφαση στο Πανεπιστήμιο της Μεσογείου που βέβαια δίνει μια μεγαλύτερη ορατότητα σε αυτές τις μορφές συνεργασίας αλλά δεν μπορεί από μόνο του να επισκιάσει τη σημαντική πρόοδο και άλλων πανεπιστημίων της περιοχής. Όλα αυτά λοιπόν έχουν σαν στόχο να δημιουργήσουμε ένα χώρο ε, δημιουργικό συνεργασία σε ανθρώπινο επίπεδο. Προφανώς η συντομία αυτής της γνωμοδότησης δεν επιτρέπει την πλήρη ανάπτυξη των ιδεών μου, αλλά περιμένω τις προτάσεις και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα συμβάλλετε όλοι επικοδομητικά στην ανάπτυξη αυτού του σχεδίου γνωμοδότησης. Ε, επίσης, η Επιτροπή Πολιτισμού έχει το, και το συναδελφό μου Φρανσουά Αλφονσί, που είναι νέο μέλος της Επιτροπής ε, <clears throat> Πολιτισμού. Δυστυχώς είναι άρθρο σήμερα, αλλά είναι εισηγητή στην, στην Επιτροπή περιφερειών και επομένως έχει να συμβάλλει τα μάλλα στην προβληματική για τις μακροπεριφέρειες. Σα ευχαριστώ, Λεκή Πρόεδρος. Ο κύριος Κουρίγια. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να σας συγχαρώ και σας προσωπικά και τους αντιπρόεδρους για την επανεκλογή σας. Άκουσα με προσοχή την παρουσίαση της συναδέλφου. Αυτή τη στιγμή έως τις προάλλες συμμετείχα και σε εργασίες Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης που είναι η αρμόδια επιτροπή για αυτό το φάκελο. Ξεκίνησε να πω στους κόλπους της Επιτροπής και μια σχετική συζήτηση. Σχετικά με το πόσες περιφέρειες χρειαζόμαστε στη Μεσόγειο. Ξέρετε, ήδη έχει ξεκινήσει η σχετική διαδικασία για την σύσταση της μακροπεριφέρειας της Αδριατικής και του Ιωνίου Πελάγους, δηλαδή για την Ανατολική Μεσόγειο ουσιαστικά. Οπότε θα θέλαμε να κατανοήσουμε καλύτερα κατά πόσον χρειάζεται να δημιουργήσουμε και μια δεύτερη μακροπεριφέρεια για τη Μεσόγειο, για τη Δυτική Μεσόγειο ή τελικά να δημιουργήσουμε μια ενιαία μακροπεριφέρεια για τη Μεσόγειο. Υπ' αυτή την έννοια Σκόπιμο θα ήταν και η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας να τοποθετηθεί για το ζήτημα αυτό. Φαντάζομαι ότι η συνάδελφος, ε, ε, η συγγήτρια θα έχει άποψη επί του θέματος και ίσως θα μπορούσαμε να υποβάλουμε και κάποιες τροπολογίες προς την κατεύθυνση. Χρειάζεται όμως να το συζητήσουμε, να εμβαθύνουμε επί του θέματος ε, εδώ στην Επιτροπή. Διότι πράγματι η Μεσόγειος είναι μια πολύ σημαντική γεωγραφική περιφέρεια και εγώ συμμερίζομαι αυτές τις θέσεις που εκφράσατε. Επίσης είναι και πηγή ε, πολιτισμού, είναι ένα στοιχείο, αν θέλετε, πηγή ταυτότητας ε, για όλους τους λαούς που μοιράζονται αυτή την θάλασσα. Αναφέρομαι βεβαίως και στην νότια πλευρά της ε, Μεσογείου, αναφέρομαι και στην Τουρκία κτλ. Ρώτω, λοιπόν πρώτα απ' όλα, προ τα πού θέλουμε να κινηθούμε. Δύο μακροπεριφέρειες για τη Μεσόγειο ή μία ενιαία μακροπεριφέρεια. Ενιαία μακροπεριφέρεια. Ε, ε, Επιτρέψτε μου και μία ερώτηση να θέσω και εγώ στην εισηγητρία. Κατανοώ το θέμα είναι σύνθετο. Αλλά ρωτώ, υπάρχουν υπάρχει κάποια δυνατότητα διαβούλευσης με αυτές τις τρίτες χώρες που θα έπρεπε να εμπλακούν σε αυτή τη συζήτηση. Αν κατάλαβα καλά, μιλούμε για την μακροπεριφέρεια της Μεσογείου, ουσιαστικά όμως της Δυτικής Μεσογείου όπου υπάρχει αν θέλετε και μια γλωσσική ενότητα που μας βοηθά, διότι οι πιο πολλές από αυτές τις χώρες μιλούν τη γαλλική. Ξέρετε όμως, επειδή εγώ συμμετέχω στην Eurolat, εντάξει, άσχετο αυτό, αλλά ε, ε, ε, η Euromed δεν είναι κάτι παρόμοιο με την Eurolat. Έτσι δεν είναι. Ρωτώ λοιπόν, πώς φανταζόμαστε εμείς αυτή τη, αυτό το θέμα. Θα είναι μια διαπολιτισμική συζήτηση και πώς θα γίνει όμως και με τα τρίτα αυτά κράτη. Ευχαριστώ. Κυρία Σάντζο Σμίτ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα. Ε, είμαι μέλος της Επιτροπής Περιφερειών και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό το ζήτημα. Το σύστημα εντός ελικών αυτών των μακροπεριφερειών είναι αρκετά θετικό και αυτό θα βοηθήσει τον συντονισμό πολλών διαφορετικών ε, ευρωπαϊκών στρατηγικών. Ε, δεν θα επιφέρει επιπλέον χρηματοδότηση αυτή η μακροπεριφέρεια. Ουσιαστικά ε, μιλάμε για, την, για κοινέ προβληματικές και έχουμε αυτό το, αυτούς τους δύο πόλους Ουσιαστικά όμως θέλουμε ε, να συγκεντρώσουμε διάφορετικούς ε, πόρους, είτε πρόκειται για διαφορετικά μία, τα ταμεία συνοχής ε, κτλ. γύρω από, τα, από, τα, από τους ίδιους στόχους. Και πράγματι, πέρα από τα προγράμματα υποδομών και όλα αυτά, καλύτερο είναι να εστιαστούμε περισσότερο στους, στην ανθρώπινη διάσταση, να μιλήσουμε για τον πολιτισμό, για την ε, παιδεία. Η ε, κυρία ε, η μίλησε για την πολιτική καλής γειτονίας. Είναι πολύ καλό αυτό να το εξετάσουμε, αυτή την πολιτική στο πλαίσιο των μακροπεφεριών μαζί με τον τέταρτο πυλώνα που μιλά για αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ, Πρόεδρε, για την επανακλογή σας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Συγήτρια. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλά δομημένη έκθεση. Εγώ δεν είμαι μέλος της ε, Επιτροπής Ρέτζη και ενδεχομένως να μην ε, γνωρίζω και πολλά πράγματα, αλλά όταν μιλάμε για την πολυπολιτισμικότητα, την περιφερειακή συνεργασία και όλα αυτά, πρέπει να εστιάζουμε και σε άλλες ε, περιφέρειες. παράδειγμα, στην Ανατολική Ευρώπη, η πολιτική καλής γειτονίας είναι μια καλή βάση πάνω στην οποία μπορούμε να οικοδομήσουμε και δεν πρέπει να ξεχνούμε αυτή την περιφέρεια. Θα πρέπει να, υπάρχει μια προσπάθεια διασύνδεσης ε, των προγραμμάτων μας με την ε, πολιτική καλής βιοτονίας και στις ε, χώρες που βρίσκονται στην Μεσόγειο αλλά και στην Κεντρική Ευρώπη για να μπορούν οι νέοι να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα που μπορούν να τους ωφελήσουν και να τα αξιοποιούν γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη των περιφερειών. Θα ήθελα πω στην κυρία Νεβεντένεβα. Σήμερα μιλάμε για τις περιοχές της Μεσογείου. Και αυτό είναι απόρρια του λεγόμενου, της λεγόμενης αραβικής άνοιξης, η οποία έγινε και ένα θερμό καλοκαίρι στη συνέχεια. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε ώστε να τον ταχύτερο με τα εργαλεία που έχουμε στον πολιτιστικό τομέα, στον εκπαιδευτικό τομέα να είμαστε και να βοηθήσουμε και αυτή την περιοχή. Δεν πρόκειται λοιπόν μόνο για θέματα χρηματικά και κονδυλίων. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε νέους ε, φορείς, νέες δομέ. Θα πρέπει απλώς να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να κάνουμε και για τις χώρες της Ανατολικής ε, Ευρώπης μέσα στα πλαίσια της πολιτικής γειτονίας. Είναι απαραίτητο όμω να δώσουμε και την απαραίτητη έμφαση στι χώρε τη νότια όχθη τη Μεσογείου, γιατί προσδοκούν βοήθεια από εμά. Εάν δεν τι βοηθήσουμε, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε καμιά δυνατότητα να τις βοηθήσουμε να πραγματοποιήσουμε αυτά τα οποία στην πραγματικότητα θέλαν να κάνουν με τις επαναστάσεις αυτές. Ο στόχος λοιπόν είναι πώς να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι ότι εμείς θα επιβάλλουμε μια κατεύθυνση σε αυτούς τους λαούς. Θα πρέπει όμως να υπάρχει μια συνεργασία και μια ανταλλαγή αμοιβαία. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που το θέμα αυτό θα αντιμετωπιστεί και στην Επιτροπή Περιφερειακών Θεμάτων. Υπάρχει κάποιος από την Κομισιόν που θα... Όχι, εντάξει, καλά, δεν, είναι τραγικό, δεν χάλασε ο κόσμος. 31 Ιανουαρίου λοιπόν, κυρία Μπεναράπ, θέλετε να πείτε κάτι ακόμα. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την σημασία που επέχει το να μην είμαι μόνη μου και να συνεργαστώ με άλλους. Αναφέρθηκε το θέμα της ε, Ευρωλάτ, της ε, Επιτροπής Συνεργασίας με την ε, Λατινική Αμερική. Εγώ είμαι και μέλος της Επιτροπής για τη Μεσόγειο, τη Ευρωμέτ και επομένω είναι πολύ σημαντική αυτή η δυνατότητα συνεργασία. Είτε έχουμε ένα πόλο ή δύο πόλου δεν έχει μεγάλη σημασία. Σημασία έχει η συνεργασία. Με δύο πόλου τα πράγματα είναι πιο ε, λογικό ίσω, αλλά εγώ νομίζω ότι θα πρέπει. Θυμίσουμε ότι οι στοχαστές ήδη από το 15ο αιώνα είχαν στο μυαλό τους μια Μεσόγειο που περιλαμβάνει και την τωρινή Κροατία το σχέδιο αυτό του Ευρωμεσογειακού Πανεπιστημίου πόσο έχει προχωρήσει. Ακούω συνέχεια, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται. Υπάρχει μια ομάδα εργασία χωρί μικρόφωνο, λέει η κυρία Μπεναρά. Με επικεφαλιστή κυρία Κράτσα μέχρι στιγμή. Είναι αυτό το πανεπιστήμιο λοιπόν το οποίο υπάρχει στην ε, Σλοβενία, αλλά υπάρχει και ένα αντίστοιχο σχέδιο στο Μαρόκο, στο ΦΕΣ, το οποίο προωθείται πιστεύω ότι θα οδηγηθούμε σε ένα δίκτυο ευρωμεσογειακών πανεπιστημίων σε όλη τη Μεσόγειο. Είναι πιο λογικό αυτό, εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρο. 31 Ιανουαρίου είναι καταληκτική ημερομηνία και μπορούμε να κλείσουμε την σημερινή μας εργασία. Τώρα έχουμε τη συνάντηση των συντονιστών. Όσοι δεν ανήκουν σε αυτό τον εκλεκτό κύκλο μπορούν να πάνε να πιούν καφέ εκτός της αιθούσης.